Dear colleagues, please. We start the explanation of votes. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Αρίας Εσεβέρια θα πάρει το λόγο ο κύριος Μεσάρος για να εξηγήσει την ψήφο του. Mr. Colleague, Mr. Μεσάρος. Mr. Μεσάρος, you have the floor.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 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο υπάρχουν ελλείψεις, ε, κυρίως στο ε, διασυνοριακό εμπόριο. Ε, δεν υπάρχουν ενιαίες εθνικές ρυθμίσεις, δεν υπάρχουν ενιαίες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Υπάρχει διαφοροποίηση των ρυθμίσεων. Διακο... Μα μίλησε, τα είπε. A határon átnyúló vásárlások 60%-ig sikertelennek bizonyul. Το 60% στην Ευρώπη έχουμε 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Δυστυχώς όμως αυτό δεν εμφανίζεται πουθενά ούτε στο διαδίκτυο. Πρέπει λοιπόν να επιτύχουμε την ενιαία ηλεκτρονική αγορά και μέσα από το διαδίκτυο. Μέχρι να βιάσει η αίθουσα από αυτούς που δεν ενδιαφέρονται. Yes. You can start. Quietly, please. <clears throat> Okay. Köszönöm, elnök asszony. <clears throat> Napjainkban már az e-kereskedelem, az internet szerves része... Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι, αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο του εμπορίου, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις, κυρίως στο διασυνοριακό εμπόριο. Δεν υπάρχουν ενιαίοι κανόνες, και δεν υπάρχουν ενιαίοι εθνικοί κανόνες κυρίως. Το 2009 κάθε τρίτος Ευρωπαίος καταναλωτής αγόρασε κάτι ηλεκτρονικά, όμως μόνο το 7% αγόρασαν από άλλο κράτος μέλος. Και έχουμε και άλλα στατιστικά δεδομένα που δείχνουν ότι περίπου το 60% των διασυνοριακών αγορών δεν μπόρεσαν να λάβουν χώρα γιατί οι πολιτές ε, δεν ε, διέθεσαν τα προϊόντα τους. Στην Ευρώπη λοιπόν υπάρχουν εμπόδια ε, στις αγορές και στο εμπόριο. Πρέπει να έχουμε μια ενιαία ηλεκτρονική αγορά, γι' αυτό και εγώ στήριξα αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μεζάρος. Για το ίδιο θέμα ο κύριος Καμάλ Σαγέντ έχει το λόγο. Mr. please. You have the floor. Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να εξηγήσω την ψήφο μου. Είναι πολύ σημαντικό, συμφωνούμε νομίζω, ότι υπάρχουν ακόμη πάρα πολλοί φραγμοί και το σημαντικό θα ήταν να μπορούμε να αγοράζουμε αγαθά και ψηφιακά και άλλου είδους από το Ιντερνετ χωρίς αυτούς τους φραγμούς. Γιατί το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι παγκόσμιο και δεν πρέπει να το περιορίζουμε μόνο στην Ευρώπη. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων δικαιοδοσιών για να αρθούν οι φραγμοί, ώστε οι πολίτες και των δύο φύλων στην Ένωση να μπορούν να αγοράζουν με τις φθηνότερες τιμές και αγαθά και υπηρεσίες από τον υπόλοιπο κόσμο μέσω του ίντερνετ. Πρέπει βέβαια να αναγνωρίσουμε ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα οι τιμές θα τείνουν να χαμηλώσουν προς το μηδέν τελικά. Παρακαλώ τους συναδέλφους να φύγουν ήσυχα από την αίθουσα όσοι δεν ενδιαφέρονται. Ο επόμενος ομιλητής ο κύριος Χανάν για την ίδια έκθεση. Ένα λεπτό παρακαλώ. One minute, Mr. Χανάν. Madam Deputy Ευχαριστώ. Ακούσαμε όλες τις κοινοτοπίες που συνηθίζονται στις οδηγίες πόσο σημαντικό είναι το Ιντερνετ δηλαδή το 2020 για να μπορέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι κτλ. Αλλά αυτό δεν διευκολύνει πράγματι το εμπόριο και τις ελεύθερες συναλλαγές. Δεν χρειάζονται οδηγίες για να μπορούν οι επιχειρήσεις να αγοραπολούν. Αυτό κάνουν ούτως ή άλλως. Εμένα ένας από τους εκλογείς μου πουλάει προϊόντα μέσω του ίντερνετ στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Αυστραλία και δεν χρειάζεται για να το πράξει αυτό ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μάλιστα χωρίς την νομοθεσία αυτή είχε λιγότερα προβλήματα. Πράγμα το οποίο εξηγεί ίσως γιατί από τότε που είμαστε μέλη της Ένωσης έχουμε πάρα πολλές εμπορικές σχέσεις με ολόκληρο τον κόσμο εκτός από τις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης. της κυρίας Σεβάρια και ερχόμαστε τώρα στην έκθεση της κυρίας Ντεβεράκα. Ο κύριος Μιλάνα έχει ζητήσει το λόγο. Mr. Milana, where is Mr. Milana? No, δεν φαίνεται να είναι στην αίθουσα. Ε, και το λόγο θα πάρει ο κύριος Αντωνιώζη. Ένα λεπτό παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως προκύπτει με σαφήνεια από την έκθεση αυτή, εδώ και πολλά χρόνια η αεροπορική κυκλοφορία αυξάνεται και παρά τις πρόοδους που έχουμε κάνει σε θέματα ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών υπάρχει παρόλα αυτά κίνδυνος ατυχημάτων. Η ισχύουσα νομοθεσία σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων είναι ουσιαστικά μία παλιά οδηγία του 1994. Ενώ ε, δεν είχαμε ακόμη τότε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αεροπορικής Ασφάλειας. Συμφωνώ απόλυτα με τη φιλοδοξία της ε, κυρίας Δεβέρακ να καταρτιστεί ένας νέος κανονισμός και να προβλεφθεί ένα νομικό πλαίσιο που θα εκχωρεί στην ΙΑΣΑ το βασικό ρόλο για θέματα ασφάλειας των ε, ευρωπαϊκών αεροπορικών μεταφορών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο κανονισμό ε, βελτιώνει τα θέματα διερεύνησης και πρόληψης των ε, αεροπορικών ατυχημάτων και χάρη στο δίκτυο και την προσοχή που δίνουμε στου συγγενείς των θυμάτων έχουμε σημαντική πρόοδο. Δυστυχώ δύο θέματα παραλείπτονται. Καταρχήν ε, η έννοια τη κουλτούρα τη ισότητα, ώστε το προσωπικό να μην βλάπτεται από αποφάσεις που λαμβάνονται ερήμοι τους και φυσικά σε καμία περίπτωση να γίνονται δεκτές κάποιες εσκεμμένες ή ε, αμελής πράξης. Επίσης δεν επιτρέπεται η συγκάλυψη πληροφοριών αλλά ούτε και η διαρροή πληροφοριών μπορεί να βλάψουν τους συγγενείς στον τύπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ισχύον σύστημα για την ε, διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων δεν είναι και πολύ αποτελεσματικό γιατί αυξάνονται οι αερομεταφορές και πυκνώνουν όλο και περισσότερο και αυτό χρειαζόμαστε έναν κανονισμό για να βελτιώσουμε την πρόληψη και τη διερεύνηση σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος. Η πρόταση για την ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Αεροπορική Ασφάλεια, του ΙΑΣΑ, που ζητήθηκε το 2002, θα βελτιώσει την διερεύνηση αυτή, αλλά χρειαζόμαστε και ένα σύστημα ευρωπαϊκών αρχών που θα επικοινωνούν μεταξύ τους και θα εξασφαλίζουν την πρόσβαση στους ε, καταλόγους επιβατών για τις διάφορες πτήσεις. Η Τσεχία συμφώνησε με το συμβασμό στο Συμβούλιο. Η έκθεση είναι πολύ τεχνική και θα βελτιώσει την ασφάλεια σε αερομεταφορές. Λιμπεράτσκι, επεξήγηση ψήφου. Έχετε το λόγο κύριε συνάδελφε για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ηφαιστειακή τέφρα δημιούργησε τεράστια προβλήματα αεροπορικών μεταφορών και είδαμε πόσο εξαρτημένοι είμαστε από αυτό το μέσο μεταφορά. γιατί η εναλλακτική λύση δεν υπάρχει. Είναι αναντικατάστατε οι αερομεταφορές, γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό το θέμα τη ασφάλεια του. Και η διερεύνηση και πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για αποτελεσματική ε, διαλεύκανση των διαφόρων περιστατικών για να αποδοθούν ευθύνε, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι η πρόληψη τέτοιων αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων. Είχαμε περιπτώσεις near collision, παρολίγο συγκρούσεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για την ασφάλεια των αεροτομεταφορών. Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για την πολύ αξιολόγηση έκθεση της κυρίας Δεβεϊράκ και να επενέσω και τους κοιοδησηγητές γιατί είναι πολύ περίπλοκο το θέμα και με ιδιαίτερη ευθύνη και επαγγελματισμό το αντιμετώπισε η κυρία Ντεφύρα. Και αυτό άλλωστε και υποστήριξε την έκθεσή τη. Σα ευχαριστώ πολύ. Τώρα ερχόμαστε στην έκθεση του κυρίου Βιντάλ Κουάντρα. Έχουν ζητήσει επτά συνάδελφοι το λόγο. Να είστε σύντομοι, σα παρακαλώ. Ο κύριο Αντωνιώζη πρώτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια πολλά κράτη-μέλη ε, υπέστησαν ε, ε, συχνά διακοπές ε, ανεφοδιασμού με αέριο. Επειδή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται όλο και περισσότερο από τον εξωτερικό εφοδιασμό, η ενέργεια ε, μπορεί να υποστεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει σε οικονομικές ζημιές στα κράτη-μέλη. Η ιδέα λοιπόν ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι καθοριστική σημασία, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το λάβουμε όλοι μας υπόψη τα χέγγια για την ε, διατήρηση του απρόσκοπτου εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μέριο κυρίως σε περιόδους κρίσης αυτό πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένας στρατηγικός στόχος. Γι' αυτό λοιπόν εγώ υπερψήφισα την έκθεση και ελπίζω ε, η έκθεση αυτή και αυτά που προτείνει να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν πράγμα το οποίο εύχεται και ο εισηγητής. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, η κρίση αερίου ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία τον περασμένο χειμώνα ε, οδήγησε ε, στο να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί ως Ευρωπαίοι. Γνωρίζουμε πολύ καλά ε, πόσο πολύ εξαρτώμεθα από τον εφοδιασμό με αέριο. Η Ευρώπη λοιπόν ε, πρέπει να αναζητήσει νέες δυνατότητες ασφάλειας στην περίπτωση που διακόπτεται αυτός ο εφοδιασμός. Εγώ συμφωνώ με τον εισηγητή ότι αν θέλουμε να διασφαλίσουμε τον απρόσκοπτο εφοδιασμό μιας παραμεθόριας απομακρυσμένης περιοχής, πρέπει να υπάρχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο σωστός μηχανισμός, ο οποίος θα λειτουργεί και σε περιφερειακό επίπεδο. Κυρία Πρόεδρε, το θέμα της ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο είναι νευραλγικό σημείο της ε, παγκόσμιας πολιτικής κατάστασης. Αλλά πάνω απ' όλα ενδιαφέρει τους ε, πολίτες, γιατί για αυτούς πάνω απ' όλα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τον ανεφοδιασμό με αυτή την πρώτη ύλη, το αέριο. Είμαι υπέρ ε, της έκθεσης, καθώς και του προσδιορισμού της ε, έκτακτης ανάγκης. Επίσης, θα πρέπει να προσέξουμε και τη γεωργική κατανομή αλλά και το κατόφλι πέραν το οποίο επιτρέπεται η παρέμβαση, το θέμα της αποκέντρωσης της προστασίας των δεδομένων, η πρόσβαση σε εμπορικά στοιχεία και φυσικά η βελτίωση της ασφάλειας ε, και της πρόσβασης στο αέριο. Πολλές ε, οικονομίες στηρίζονται στην οικονομία με αέριο, γι' αυτό και εγώ υπερψήφισα την έκθεση που την έκανα πολύ σωστή. Εγκρίναμε πολύ σημαντική έκθεση για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο. Προτείνονται πολύ σημαντικά και πολύ σωστά μέτρα. Βέβαια δεν εξασφαλίζουν απόλυτη ασφάλεια στην κοινωνία και στην οικονομία σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό με αέριο. Τα συμβάντα των τελευταίων χρόνων έδειξαν ότι οι δραστηριότητες πολλές χωρών μελών ε, καθορίζονται κυρίως από τα δικά του συμφέροντα και όχι από την ε, φιλοδοξία δημιουργίας μιας αλληλέγγυας ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να εξαρθρώσουμε τα μονοπόλια, θα πρέπει να, να συνδυάσουμε την ε, πολιτική στο αέριο με τη διεθνή πολιτική. Χρειαζόμαστε υποδομές. Επίσης, Χρειαζόμαστε κάποιες κοινέ ε, υπερεθνικές δράσεις. Όλες αυτές είναι δραστηριότητες που θα πρέπει να υλοποιηθούν για την ε, πραγματοποίηση μιας ευρωπαϊκής τέτοιας πολιτικής ασφάλειας. Η ε, έκθεση αυτή μας προτείνει τα πρώτα βήματα για την οικοδόμηση μιας τέτοιας πολιτικής. Κυρία Πρόεδρε, η ε, ασφάλεια των προμηθειών μας ε, αέριο είναι κάτι από τους πιο σημαντικούς τομείς της ενεργειακής ασφαλείας και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μιλήσουμε για αυτό το θέμα με μια φωνή από τους σημαντικότερους στόχους. Εκτιμώ ιδιαίτερα την εργασία λοιπόν του κυρίου Ότιγκερ αλλά θα ήθελα να πω ότι μετά από πενταετή συζήτηση πενταετή συζήτηση είναι κάτι το υπερβολικό Πρέπει να διαφοροποιηθούν οι ενεργειακές μας πηγές διότι η Ρωσία χρησιμοποιεί, εκμεταλλεύεται το μονοπόλιο της για να ασκήσει πολιτικές πιέσεις επί των βαλτικών παραδείγματος χάρη χωρών. Πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή της αλληλεγγύης που είναι μία από τις βάσεις της ενωσιακής πολιτικής. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια κατάσταση όπου όλο το αέριο μεταφέρε, που μεταφέρεται προς την Ευρώπη προέρχεται από τη Ρωσία. Πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας με τις χώρες του Καυκάσου και να έχουμε εναλλακτικέ πηγές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ υπερψήφισα αυτή τη ε, διάταξη. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητο να έχει ξεκάθαρες ε, ρυθμίσεις όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό. Η περσινή διαμάχη κατέδειξε πόσο μεγάλη είναι η εξάρτησή μας από ενέργεια που προέρχεται από τρίτες χώρες. Αυτή λοιπόν η ρύθμιση επιτέλους αντιμετωπίζει το πρόβλημα για να προλάβουμε το ενδεχόμενο μελλοντικών κρίσεων. Σημαντικό βήμα προς τα εμπρό. Τα κρατη καλούνται να ε, εγγυώνται και αυτά τον εφοδιασμό με τις απαραίτητες δομές και τις απαραίτητες υπηρεσίες. Επίσης καλούνται να έχουν και ε, προγράμματα έκτακτης ανάγκης. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό φτάνουμε στην εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας που είναι τόσο σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη δική μου την πολιτική ομάδα. Ε, το, η ρύθμιση 62 αναφέρεται σε αυτό όλα αυτά. Επίσης, ε, η χώρα μου ε, θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε διορατικοί, να έχουμε ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας ε, με όσους διαθέτουν μεγάλες ποσότητες αερίου. Καλό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σήμερα εγκρίναμε τον κανονισμό για την ασφάλεια των προμηθειών μας σε αέριο που είναι σημαντική πρόοδος στο δρόμο της εφαρμογής της ενεργειακής μας πολιτικής και αποτελεί επίσης πρόοδο και ως προς την περιφερειακή συνεργασία και αλληλεγγύη. Εγώ υπερψήφισα διότι αναμένω ο κανονισμός αυτός να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν απομονωμένες περιοχές της Ένωσης ως προς την ενέργεια όπως οι βαλτικές χώρες. Επίσης πιστεύω ότι θα δοθεί έτσι μια όθηση για την εφαρμογή διάφορων ανεφάρμοστων μέχρι τώρα προγραμμάτων. Ο κανονισμός βέβαια έχει και ορισμένες ελλείψεις, όπως την κατάργηση της ιδέας να περιοριστούν τα μονοπόλια όπως της Gazprom και δεύτερον την περιβαλλοντολογική προστασία. Ελπίζω κάποτε η Κομισιόν να αρχίσει να εφαρμόζει και το εργαλείο αυτό για την, το περιβάλλον. Για τη Συμφωνία Επενδυσδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακιστάν τέσσερα, τέσσερες αιτήσεις προσωπικής έχουμε. Ξεκινάμε από τον κύριο Μαστέλα. Ευχαριστώ ε, Πρόεδρε. Αυτή η συμφωνία έχει ως στόχο να διευκολύνει τις διοικήσεις των κρατών μελών έτσι ώστε να ε, είναι πολύ πιο εύκολη η επαναπομπή. Να υπάρχουν όλες οι τεχνικές ρυθμίσεις, ε, να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Εγώ λοιπόν υπερψήφισα γιατί είμαι πεπισμένη ότι αυτή η συμφωνία είναι πολύ απαραίτητη. Είναι θεμελιώδε εργαλείο στον αγώνα κατά τη λαθρομετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία περιλαμβάνει ε, και άλλε ρυθμίσει. Τα κράτη-μέλη καλούνται να σέβονται το διεθνές δίκαιο και ε, την περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να υπάρξει επαναπομπή ή επανεισδοχή από την άλλη πλευρά να ρυθμίσει το θέμα από τα εθνικά δικαστήρια. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ε, ε, λαμβάνεται η επανεισοχη απο την αλλη πλευρα να ρυθμισει το θεμα απο τα εθνικα δικαστηρια γι αυτο λοιπον θα πρεπει να λαμβανεται η χωρα και η δυνατότητα άμεσης ε, επαναπομπής. Έχουμε λοιπόν μια μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί από το θέμα και θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι δυστυχώ το Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει από την Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει λοιπόν να μα ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. έχει το λόγο ε, how Τραγική ηρωνία η Ένωση σήμερα το Κοινοβούλιο εγκρίνει την έκδοση, την εκδίωξη πτωχών Πακιστανών εκτός Ένωσης σε μια χώρα όπου θα αντιμετωπίσουν ακόμη περισσότερα προβλήματα. Οι αγρότες και οι εργάτες του Πακιστάν υποφέρουν περισσότερο παρά ποτέ από τις πλημμύρες. Έχουν καταστραφεί σωτιές, ε, πεθαίνουν τα κοπάδια και εκατομμύρια, πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι αφορούνται από αυτό. Καλύτερα θα κάναμε να καταπολεμήσουμε την ανέχεια στο Πακιστάν ή να ακυρώσουμε τη χρέωσή του και τα χρέη των πτωχών αγροτών ή να αυξήσουμε τη βοήθεια που μπορούμε να χορηγήσουμε όχι βέβαια μέσω της διεφθαρμένης κυβέρνησης αλλά με δημοκρατικό έλεγχο των εργατών και αγροτών. Αυτά όλα θα ήταν πολύ καταλληλότερα μέτρα από τον κανονισμό αυτόν. Ένα λεπτό επίσης σε ό,τι αφορά τη συμφωνία πανεισδοχής με το Πακιστάν. Φαίνεται ότι διευρύνεται η δυνατότητα των χωρών μελών να επαναπατρίσουν λαθρομετανάστες προς το Πακιστάν. Και αυτό θα ήταν ευκταίο για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά καλύτερα να αποφασίζει μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο ως κυρίαρχο κράτος ποιους θα επαναπατρίζει και ποιοι όχι. Γιατί αν ψηφίσουμε υπέρ μιας τέτοιας έκθεσης είναι σαν να εκχωρούμε ένα τέτοιο δικαίωμα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρμόδια να ελέγχει το θέμα της μετανάστευσης, της λάθρο μετανάστευσης. Κάθε χώρα είναι κυρίαρχη και θα πρέπει να το αναλάβει μόνη της. Και ζητήσει το λόγο, αλλά δεν φαίνεται στην αίθουσα. Οπότε ερχόμαστε στην επόμενη έκθεση, έκθεση Καζάκ, εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία. Μάλλον. Παντού. I'm sorry, I was sitting. Λυπάμαι, ήμουν σε λάθος κάθισμα. Δεν θέλω να πω ότι οι φιλελεύθεροι είναι της Δανία είναι ικανοποιημένη από τη Συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Πακιστάν. Και επιτέλου, μετά από πολλά χρόνια διαπραγματεύσεων ε, ανάμεσα στο Πακιστάν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήξαμε σε συμφωνία που θα επιτρέψει την επανεισδοχή μεταναστών που δεν πληρούν πλέον τι προποθέσει ε, για την είσοδο ή παραμονή διαμονή στα κράτη-μέλη. Η συμφωνία αυτή είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα γιατί το Πακιστάν είναι μια πολύ σημαντική χώρα προέλευσης αλλά και ε, διέλευσης μεταναστών. Με τη συμφωνία αυτή το Πακιστάν ε, αναλαμβάνει να ε, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ξαναδεχθεί τους υπηκόους της, κάτι που θα βελτιώσει και θα αυξήσει την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Ε, τώρα για την επόμενη έκθεση Καζάκ, όπως είπα εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία, έχουν ζητήσει το λόγο οκτώ συνάδελφοι. Προσπαθήστε να μην ξεπεράσετε το ένα λεπτό ο καθένας. Η κυρία Μουσκαρντίνη θα πάρει πρώτο λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ είμαι υπέρ της έκθεσης Καζάκ για τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία όπως ψηφίστηκε η έκθεση αυτή ε, στην Ολομέλεια. Η ε, Τουρκία... Στην Τουρκία εξακολουθεί να υπάρχουν ε, πάρα πολλά εμπόδια κυρίως εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αν θέλουμε λοιπόν να συμβάλλουμε στην εξέλιξη των εμπορικών σχέσεων, η Τουρκία πρέπει να λάβει υπόψη στη θέση αυτού του κοινοβουλίου. Δηλαδή ε, να δεχθεί το κοινωτικό κεκτημένο όσον αφορά τις εμπορικές ανταλλογές. Ε, να καταπολεμήσει την παραποίηση και να μην ξεχνάει ότι υπάρχουν τομείς όπως ο φαρμακευτικός όπου υπάρχει η εγγύηση ελεύθερης διακίνησης των φαρμάκων και αν δεν γίνεται αυτό ε, ε, προβλέπονται σοβαρές κυρώσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει η Τουρκία να αποφύγει διακριτική μεταχείριση έναντι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ε, κυρίως σε κρατικούς διαγωνισμούς και σε κρατικές προμήθειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Φυσικά και καταψήφισα την έκθεση Καζάκ γιατί είχα εκθέσει και τα επιχειρήματά μου ως προς την μεροληψία του. Δεν μπορώ να υπερψηφίσω μια έκθεση όταν ε, ο εισηγητής σπούδασε με χρηματοδότηση της τουρκικής κυβέρνησης. Υπάρχει ασυμβίβαστο κατά τη γνώμη μου. Σύγκρουση συμφερόντων. Δεν νομίζω ότι είναι αντικειμενικό ο κύριο Καζάκ στην έκθεσή του, γι' αυτό και δεν μπορώ να τον υποστηρίξω. Ορισμένα σημεία και παράγραφοι της έκθεσης είναι τελείως άσχετα με το εμπόριο και την οικονομία. Απλώς περιέχουν εγκόμια προς την τουρκική κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που έκανε, για τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Ναι, είναι αλήθεια ότι ο στρατός και το δικαστικό σύστημα εξασφάλισαν τον κοσμικό χαρακτήρα της Τουρκίας, αλλά όσο προχωράμε τόσο περισσότερο ε, οδεύει προς τον ε, θρησκευτικό ισλαμικό χαρακτήρα η Τουρκία. Δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ μιας τέτοιας έκθεσης. Eh, Κύριε Πρόεδρε, ο ρόλος ε, της Τουρκίας ε, με στη σχέση με την Ευρώπη και στον παγκόσμιο χαρτί ε, επεκτάθηκε τα τελευταία χρόνια γιατί εκμεταλλεύεται τη γεωπολιτική της θέση. Η υλοποίηση λοιπόν τελειονικής ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1996 επέτρεψε να βελτιωθούν οι εμπορικές ανταλλαγές και οι οικονομικές σχέσεις κυρίως αναφορά την ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων. Τελευταία χρόνια έχει γίνει ε, μια μεγάλη, ένα μεγάλο βήμα προ τα εμπρό ε, με τον τελωνιακό κώδικα και το σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι τελευταία χρόνια η Τουρκία έχει γίνει ε, σημαντικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στον πέμπτο, στην πέμπτη θέση για τι εξαγωγέ. Έχουν γίνει αρκετέ επενδύσει των Ευρωπαίων, κυρίω σε τομεί που προσφέρουν υπεραξία. Πρέπει σας πω ότι συμφωνώ ότι θα πρέπει ο τομέας των, ε, ο τελωνιακός τομέας, τομέας να λειτουργεί πολύ καλύτερα. Frau Präsidentin, zwischen der Europäischen Union und Κυρία Πρόεδρε, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ε, Τουρκία υπάρχουν πολλές εμπορικές σχέσεις. Ε, το 1996 συστήθηκε η Τελωνιακή Ένωση ε, και παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εμπορικά προσκόμματα. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που σήμερα το Κοινοβούλιο καλεί την Τουρκία να άρει αυτές τι δυσκολίε που έχει δημιουργήσει να εγκρίνει το σύστημα των ποσοστώσεων για τα γεωργικά προϊόντα. Επειδή αυτά, το δικό του σύστημα δεν ταυτίζεται με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από κοινού πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε τα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από την Τουρκία να απολαύουν των ίδιων προδιαγραφών που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω συμφωνήσει, αλλά θα έλεγα ακόμα υπολείπονται πολλά. Ας ξεκινήσουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μποσινιόρ. Ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για τη δουλειά του και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το επιχείρημα. Ε, παρά το γεγονός ότι συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την Τουρκία και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύσκολη στιγμή για την Ευρώπη και για την Τουρκία η Τουρκία είναι ένας πολύ καλός εμπορικός εταίρος, ε, δηλαδή έχει κάνει βήματα προς τα εμπρός ε, και είναι η φυσική πόρτα προς την Ασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας. Τα στοιχεία είναι καλά, ε, ικανοποιητικά, τέτοιου είδους εμπορικές σχέσεις πρέπει βεβαίως να βελτιωθούν έτσι περαιτέρω. Γι' αυτό λοιπόν το 16 και το 20, τα σημεία αυτά τα δέχομαι, εκεί καλείται η Τουρκία να μειώσει τα προσκόμματα για εισαγωγή, κυρίως στον φαρμακευτικό τομέα. Και τέλος, θεωρώ ότι πράγματι είναι σημαντικό να υπάρχουν καλύτερες εμπορικές σχέσεις, να βελτιωθεί το τελωνιακό θέμα έτσι ώστε να είναι και πιο υποφελείς οι ανταλλαγές. Eh, Πρόεδρε, εγώ υπερψήφισα την έκθεση Καζάκ, διότι εξέταζε το εμπόριο και τις οικονομικές πτυχές των ανταλλαγών και τρόπους βελτίωσης του ως προς τη σχέση με την Τουρκία. Απέσχον όμως επί της τροπολογίας ένα γιατί δεν νομίζω ότι η Τουρκία πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια δεν ήταν αυτό το θέμα της έκθεσης. Κατά τα υπόλοιπα την υποστηρίζω. Κυρίες και κύριοι, παρά της βελτίωση των σχέσεων μας με την Τουρκία, υπάρχουν ακόμη κάποιοι δασμολογικοί και μη δασμολογικοί δασμοί στο εμπόριό μας. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες που χρήζουν απλούστευσης προβληματικά θέματα υπάρχουν και από τις δύο πλευρές. Ε, το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας, ε, της τήρησης διαφόρων δικαιωμάτων, ε, το θέμα της παραποίησης πολλών προϊόντων είναι πολύ σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν και τις δύο πλευρές. Παρ' όλα αυτά μας ενδιαφέρει η εταιρική σχέση με την Τουρκία, αλλά θα πρέπει να δούμε ποια είναι η αιτία των εμπορικών φραγμών που ισχύουν. Επίσης, Έχουμε την μακροχρόνια προσδοκία της Τουρκίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ίσως ε, ψάχνει ε, εναλλακτικούς εταίρους ε, σε αυτή την προσπάθεια η Τουρκία. Θα πρέπει λοιπόν η ανάλυση των σχέσεών μας να γίνει και υπό το φως των πρόοδων που κάνει η Τουρκία και σε θέματα νομοθετικά. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά και ψήφισα υπέρ της έκθεσης Καζάκ και μάλλον συγγνώμη, ψήφισα υπέρ της τροπολογίας του και κατά της έκθεσης ε, Καζάκ. Μπορούμε κάλλιστα να έχουμε αγαστές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία χωρίς ε, να γίνει σώνη και καλά μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα αυτή. Υπάρχουν ε, πολλά ελλείμματα σε ό,τι αφορά τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας. Άλλωστε, το κόμμα ΑΚΠ οδήγησε μια ριζοσπαστικοποίηση της χώρας αυτής ε, και μια στροφή προς ε, πιο ριζοσπαστικό Ισλαμισμό. η εφαρμογή του συντάγματος ε, είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη διατήρηση του κοσμικού ε, κράτους στην Τουρκία και μια κυβέρνηση υπέρ της κοσμικότητας. Με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, η κυρία Ροντζούλη θα πάρει πρώτο το λόγο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Μίσης Ροντζούλη. scusi Presidente. Grazie. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα η έκθεση που εγκρίθηκε ακολουθεί την σωστή κατεύθυνση για να προστατεύσουμε την βιοπικιλότητα και τα οικοσυστήματα. Η έννοια της βιοπικιλότητας επιτέλους συνδέεται με την υπεύθυνη διαχείριση για να διαφυλάξουμε τον πλανήτη μας και για τις μελλοντικές γενιές είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή να υπάρχουν πολιτικές που διατηρούν την βιοπικιλότητα. Ο στόχος του να ε, ανασχεθεί η απόλυτη βιοπικιλότητα μέχρι το 2010 δεν επιτεύχθηκε και γι' αυτό πρέπει τα κράτη-μέλη και οι αρμόδιοι θεσμοί ε, να λάβουν τα σωστά μέτρα. Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από τον Νότο μέχρι το Βορρά ε, διαφυλάσσει την βιοπικιλότητα, μια μοναδική βιοπικιλότητα. Πρέπει λοιπόν να διαφυλάξουμε αυτή την περιβαλλοντική κληρονομιά γιατί αυτό το φίλουμε και στους εαυτούς μας και στις επόμενες γενιές. Κύριε Πρόεδρε, αυτή την έκθεση για την εφαρμογή των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την υπερψήφισα. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα δεν επιτεύχθηκαν λόγω του ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Δεν βρήκαμε τα απαραίτητα στοιχεία, η χρηματοδότηση δεν είναι ε, και δεν ε, βλέπετε ενσωμάτωση ε, στη νομοθεσία γενικότερα. Χρειαζόμαστε καλύτερες εκθέσεις, καλύτερη κάλυψη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να συμπεριφέρεται με πολιτικό τρόπο αλλά να παραμείνει επί της ουσίας. Καλούμεθα να προστατεύσουμε τη φύση και το μέλλον της ανθρωπότητας ε, και όχι τις ε, περιφέρειες των ε, κρατών μελών. Κύριος Μαστέλα, κύριε κυρία Πρόεδρε, η βιοπικιλότητα και τα οικοσυστημότητα ε, και ε, ο αγώνας διατήρησής τους, αυτός είναι ένας αγώνας για την κοινωνία μας. Το να ε, διατηρήσουμε την απώλεια της βιοπικιλότητας, αυτό είναι και ένα πολιτικό και οικονομικό στοιχείο που μας αφορά και αφορά και τις επόμενες γενιές. Με βάση την πράξη, η πορυβαλλοντική πολιτική της κοινότητας πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να έχουμε τη σωστή προσέγγιση με βάση και την αναλογικότητα και την επικουρικότητα. Όμω πολύ συχνά υπάρχουν διαφορέ στα κρατημέλη και αυτό δεν επιτρέπει μια σωστή εφαρμογή. Σωστό με την εισηγήτρια ότι η τομεακή προσέγγιση τη ευεπικοινότητας κατ' ουσίαν ευνοεί την κατάτμιση ε, και δεν ευνοεί το στόχο μα. Εάν λοιπόν αυτή η κατάτμιση και η οικονομική θέλουμε να έχει θετικό αποτέλεσμα ε, θα πρέπει να αφήσουμε αυτή την ιδέα του, της επιλεκτικής ε, προσέγγισης ε, να μην ε, παραλείπουν τα κράτη-μέλη να ε, δαπανούν τα απαραίτητα κονδύλια για τη διατήρηση της βιοπικιλότητας. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 42% των θηλαστικών και 45% των ψαριών και των πουλιών που απειλούνται με εξαφάνιση. Δυστυχώς τι συμβαίνει. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη, αυτό όμως δεν το έχουν συνειδητοποιήσει όλοι, ούτε και οι πολίτες, ούτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, όσον αφορά τους αριθμούς αυτούς, ε, κανείς δεν κάνει τίποτα. Ε, πάντως πρέπει να εφαρμόσουμε περιβαλλοντικά μέτρα και να στραφούμε κατά των παραβατών. Αν βέβαια είμαστε σοβαροί και αν επιθυμούμε στις επόμενες γενιές και στα ε, παιδιά μας ε, να δώσουμε ένα πλανήτη για να μπορούν να ζουν. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ ε, στηρίζω τα προτινόμενα μέτρα που οδηγούν στο να προλάβουμε ζημιές, μελλοντικές ζημιές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ε, βιοπικιλότητα είναι ε, καθοριστική σημασία ε, για τον αυξανόμενο πληθυσμό του πλανήτη και αποτελεί προϋπόθεση για το ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή. Αυτή η βιολογική ποικιλότητα απειλείται από τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσουμε την απώλεια της βιοπικιλότητας και να προσπαθήσουμε να άρουμε τις ζημιές. Οι καλύτερες προϋποθέσεις είναι η αηφορία, η βιωσιμότητα. Εδώ λοιπόν τα κράτη-μέλη είναι σύμμαχοι, δεν είναι εχθροί και νομίζω ότι στο μέλλον αυτή την προσέγγιση πρέπει να έχουμε. Και μία θετική είδηση. Στη δική μου την περιφέρεια ε, κατορθώσαμε στην Σαξονία να προστατεύσουμε το λύκο. Και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα και να ακολουθήσουν και άλλα. Ευχαριστώ πολύ και για την είδηση την καλή. Η κυρία Φλεσίκο Βαμπένοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για το περιβάλλον και για την ε, βιοπικιλότητα υπάρχει σήμερα ένα σημαντικό πρόβλημα ε, που είναι το επίπεδο διαβίωσής μας, η κατανάλωση ε, στην οποία καταλήγουμε εμείς και αγνοούμε την ε, βιοπικιλότητα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε ε, τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας έτσι ώστε να αποφύγουμε περαιτέρω απώλειες. Οφείλουμε να λάβουμε νέα μέτρα και να θεσπίσουμε νέους νόμους, κυρίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πολλοί πολίτες πιστεύουν ότι η απώλεια της ε, βιοπικιλότητας ε, είναι κάτι που δεν τους αφορά άμεσα. Οι πολίτες ε, δεν έχουν τις επαρκείς γνώσεις για το τι πρέπει να κάνει κανείς ε, να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Εγώ συμφωνώ με τον εισηγητή ότι πράγματι πρέπει να δρομολογήσουμε μια μεγάλη εκστρατεία. Πράγματι η βιοπικιλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για τον άνθρωπο. Εμείς όμως ε, κάνουμε τα πάντα ε, για να χάσουμε αυτό το αγαθό. Το Natura 2000 είναι ένα πρόγραμμα που ε, θα μπορούσε να μας προστατεύσει πρέπει να επιβάλλονται μεγαλύτερα πρόστιμα για ε, εταιρείε οι οποίες ε, καταστρέφουν τη βιοποικιλότητα. Εγώ στηρίζω την έκθεση Lange κυρίως στα σημεία εκείνα όπου η εισηγήτρια μιλάει για αντισταθμιστικές αποζημιώσεις ε, για τους ε, γεωργούς που αγαπούν το περιβάλλον ε, και θέλουν να το προστατεύσουν. Παρόλα αυτά χρειάζονται οι γεωργοί αυτοί την οικονομική βοήθεια γιατί δεν μπορούν να στηριχθούν στα δικά τους τα μέσα. Κουνάειτε τώρα έχει λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ασφάλιση της βιοπικιλότητας είναι θέμα που συνδέεται με πολλά άλλα την αλληλεία, τη γεωργία. Όλοι αυτοί οι τομείς επηρεάζονται από τη βιοπικιλότητα και επηρεάζουν το περιβάλλον, παραδείγματος χάρη της Βαλτικής θαλάσσης, που είναι από τις πιο μολυσμένες στην Ένωση πρέπει να φροντίσουμε τη βιοπικιλότητα. Μέχρι τώρα δεν είχαμε ασχοληθεί όσο θα έπρεπε. Η κάθε χώρα μέλος βέβαια πρέπει να κάνει και τη δική της προσπάθεια να προσπαθήσει να διατηρήσει βιώσιμη αλληλεία εφαρμογή του Natura 2000, μείωση της μόλυνσης και διάφορα άλλα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί καταλήγουν στην τρομερή μόλυνση της Βαλτικής και σε απώλεια της βιοπικιλότητάς της. Επίσης νομίζω ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε, να μειώσουμε τις ανεύθυνες δραστηριότητες πολλών βιομηχανικών τομέων. Λήψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Δύο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Ούντζας πρώτος. Ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η ψηφοφορία που έλαβε σήμερα χώρα για την έκθεση αυτή ήταν ε, ξεκάθαρη το αποτέλεσμά της ε, και καταλήγει ότι πρέπει να προλάβουμε τις οικολογικές ε, καταστροφές τα μέτρα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα μέτρα πρόληψης, αποδείχθηκε δυστυχώς ότι είναι ανεπαρκή. Ε, εφαρμόζονται εδώ και ένα χρόνο και γι' αυτό λοιπόν πλέον καταλήγουμε στο ότι είτε θα πρέπει να υπάρχουν καλύτερες παρεμβάσεις και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή να αλλάξουν οι ε, προϋποθέσεις για πρόσβαση στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Εξίσου σημαντικό είναι οι ε, περιφέρειες και οι αρμόδιοι φορείς ε, να τύχουν τις απαραίτητες σημασίες. Εδώ λοιπόν ζητώ να γίνεται καλύτερη ενσωμάτωση των φορέων αυτών στα λειτουργικά προγράμματα. Αυτό θα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, ένα από τα πολλά που κάνουμε προς την κατεύθυνση της βελτιωμένης προστασίας του περιβάλλοντος και των περιφερειών. Κύριο Σπυρίλο τώρα το λόγο έχει. Popolamento η απερίμωση και ε, οι τόσο πολλές ε, καταστροφές, ε, οι πυρκαγιές, οι ξηρασίες, όλα αυτά αναγκάζουν τα κράτη-μέλη να παρέμβουν με λίγους πόρους. Το πιο σημαντικό ερώτημα που θέτω είναι το εξής. Πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την επιβίωση του αγροτικού πληθυσμού που πολύ συχνά εκτίθεται σε θεομηνίες και αυτές οι θεομηνίες γονατίζουν τα εισοδήματά τους. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει ε, να συστήσει ένα ε, δημόσιο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας για τη γεωργία που θα μπορεί να αντιμετωπίζει τους κινδύνους, την οικονομική η αστάθεια των γεωργών μετά από φυσικές θεομηνίες, καταστροφές ανθρωπογενείς όπως ακριβώς αναφέρεται στο σημείο 37 της πρότασης του κυρίου Φεραίρα την οποία και υπερψήφισε. Η επόμενη έκθεση τώρα και η τελευταία που εξετάζουμε ε, είναι η έκθεση Θεοχάρους «Μείωση της φτώχειας και δημιουργία απασχόλησης στις αναπτυσσόμενες χώρες» Έχουν ζητήσει το λόγο έξι συνάδελφοι. Η κυρία Ροντζούλη δεν φαίνεται να είναι στην αίθουσα και πηγαίνω στον επόμενο εγγεγραμμένο συνάδελφο, τον κύριο Καλινόφσκι. Σας ευχαριστώ. Η παροχή βοήθειας στους φτωχότερους είναι από τις βασικές αρμοδιότητες ή τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό και συγχαίρω θερμά την κυρία Θεοχάρους για την έκθεσή της. Είμαι και μέρος της Επιτροπής Γεωργίας και ως Γεωργός θα ήθελα να ε, αναφερθώ στο σημείο 94 που μιλάει για την κοινή γεωργική πολιτική. Η αναθεώρηση του συστήματος ενίσχυσης είναι απαραίτητη, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε επανάληψη ε, της κατάστασης που είχαμε μετά την μεταρρύθμιση κυρίσης οργάνωση αγοράς ζάχαρης, γιατί οι φτωχότεροι παραγωγοί του των χωρών επωφελήθηκαν περισσότεροι από την ΚΟΑ, αλλά πολύ περισσότερο ε, ευνοήθηκαν όχι οι μικροκαλλιεργητές, αλλά οι μεγάλες πολυεθνικές, οι μεγαλογεοκτήμονες της ε, Αμερικής. Θα πρέπει λοιπόν να επισημάνω ότι ψήφισα κατά της παραγράφου 94, αντίστοιχα υπερψήφισα το σύνολο της έκθεσης. Έχει το λόγο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η προηγούμενη έκθεση ήταν πολύ ισορροπημένη. Παρ' όλα αυτά την καταψήφισα γιατί ακόμη και μία ισορροπημένη έκθεση ξεκινάει από το, την προϋπόθεση ότι χρειαζόμαστε ε, παροχή μεγαλύτερης ενίσχυσης προς φτωχότερες χώρες και ιδιαίτερα τις αφρικανικές χώρες και ότι έτσι θα βοηθήσουμε την Αφρική να ξεπεράσει τα προβλήματά Αυτό μπορεί να είναι πολιτικός ορθό, αλλά στην ε, πράξη δεν ισχύει. Στην Αφρική έχουμε εκατοντάδες ε, εκατομμύρια ενίσχυση που έχουμε αποστείλει ως Ευρωπαϊκή Ένωση στις αφρικανικές χώρες και αντί να μειώνεται η φτώχεια στην Ήπειρο αυτή αυξάνεται. Δεν μπορούμε να μιλούμε λοιπόν για έκτακτη ενίσχυση. Θα πρέπει να προβλέψουμε διαφορετικούς μηχανισμούς βοήθειας και να εξασφαλίσουμε παροχή της ενίσχυσης σε αυτούς που πραγματικά τη χρειάζονται. Μιλούμε για 1,8 τρισεκατομμύρια που είναι οι πραγματικέ ανάγκε της Αφρικής, αλλά είναι αδύνατο να βρούμε αυτό το πόσο για να βοηθήσουμε την Αφρικανική Ήπειρο. Κύριε Μασονιώτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για το έργο της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν ασχολείται με την στήριξη των αναπτυσσομένων χωρών και θα ήθελα ε, να πω ότι πράγματι πιστεύω ακόμα υπολείπονται πάρα πολλά. Για να βελτιωθεί η κατάσταση αυτών κρατών θα πρέπει να βελτιωθούν οι προδιαγραφές ε, στο δικαίω για την εργασία ε, και θα ήθελα κυρίως να υπογραμμίσω το ότι στηρίζω το σημείο υπαριθμών 38 όπου αναφέρεται η σημασία της ισότητας των δύο φύλων για την οικονομική επιτυχία των κρατών. Οι γυναίκες ε, πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο χώρο της εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει μέσα από όλα τα απαραίτητα εργαλεία να προσπαθήσει να ε, εκριζώσει την ε, εργασία των ανηλίκων. Αυτό το αναφέρει η συγκήτρια στο σημείο υπαριθμών 38 που αυτή τη στιγμή στο βαθμό που δεν εφαρμόζεται αυτό το μέτρο είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την εξάλληψη της φτώχειας. Εγώ λοιπόν υπερψήφισα αυτή την έκθεση. Ο κύριος Καμάλ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κανένα δεν μπορεί να είναι κατά του στόχου τη μείωση τη φτώχεια και τη δημιουργία απασχόληση στι αναπτυσσόμενε χώρε. Πήγα πριν από δύο χρόνια στην ακτή του Ελεφαντοστού και μάλιστα συνομίλησα με νέου πολιτικού από τη χώρα αυτή και του ρώτησα πώ πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να σα βοηθήσει. Μου είπαν λοιπόν, φροντίστε πρώτα απ' όλα η ενίσχυση που θα προσφέρετε δεν θα ενισχύει μόνο τι διεφθαρμένε κυβερνήσει και την δρέωσή του στην εξουσία. Αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε. Ναι. Να παταχθούν τα κρατικά μονοπόλια που προσφέρουν κακή ποιότητα υπηρεσίε. Σε ό,τι αφορά την κοινή γεωργική πολιτική, μα είπαν καταργήστε, τις, καταργήστε την και φροντίστε να ενισχύσετε περισσότερο την γεωργία και στηρίξτε κάποια ε, μέτρα στήριξης ε, που δεν θα συνιστούν όμως ένα είδος φιλοπεριβαλλοντικής ε, απεικιοκρατικής πολιτικής. Το ΕΡΚ και οι σοσιαλιστές ε, θέλουν ουσιαστικά να περιορίσουν ε, τις επενδύσεις στις χώρες αυτές. Τέτοιου είδους χαζομάρες θα πρέπει να αποφευχθούν. Κύριος τώρα έχει το λόγο. Ε, Εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή με τα χαράς για να φανεί ότι δεν ξεχνούμε όσους υποφέρουν από την ανέχεια Ιδίω μετά την οικονομική κρίση. Όταν πήγα στην Αφρική πριν από μερικά χρόνια, ε, διάβαζα στις εφημερίδες ο, πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός των αντιτιθεμένων στην δραστηριότητα των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Γιατί έλεγαν ότι έχουν ιδιωτική αντίληψη των πραγμάτων. Πρέπει λοιπόν και εμείς εδώ στη συζήτησή μας να μην βλέπουμε τα πράγματα μεμονωμένα και να έχουμε σχέσεις και με τους τοπικούς ηθήνοντες και όχι μόνο με την κεντρική κυβέρνηση και τις επίσημες ΜΚΟ. που θα ξαναξεκινήσουμε. Καλή όρεξη. Σας ευχαριστώ.